Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Βάσει του άρθρου 211 παράγραφος 3 η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων προτείνει την εξής ερμηνεία του άρθρου 51 ε, διαδικασίες σε περιπτώσεις ε, μικτών συνεδριάσεων επιτροπών. Αν ε, έχετε την διατύπωση στους φακέλους σας, αν δεν προβάλλετε ενστάσεις, ε, μέχρι να εγκριθούν τα πρακτικά θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προτείνει την εξής ε, ερμηνεία του άρθρου